ψηφίσετε. Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, Mr. Pitella Ο κύριος Πιτέλα έχει ζητήσει τον λόγο για διαδικαστικό. Τε... Πρόεδρε, συνάδελφοι, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Ήθελα να σας ζητήσω να μεταφέρετε στον πρόεδρο Ταγιάννη κάποια δημόσια δήλωση, μια καταδίκη προσωπική και θεσμική για τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον βουλευτή Κόρμπιν Μίκελ. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να γίνονται τέτοιε δηλώσει και να ακούγονται τέτοιε επονίδιστες δηλώσει κατά των θεμελιωδών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω η ισότητα των φύλων. Επ' αυτών θεμελιώνεται ολοκληρή Ένωση. Δεν μπορεί όλα αυτά να ακούγονται στον οίκο των βουλευτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να παραμένουν ατιμόρυτε τέτοιε συμπεριφορέ. Γι' αυτό ζητούμε από τον πρόεδρο Ταγιάννη να ε, λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Και εξ ονόματο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Δημοκρατών θέλω να ε, εκφράσω την σαφή μας καταδίκη και να επαναλάβω την υποστήριξή μας ε, για την ισότητα ε, ανδρών και γυναικών και την καταδίκη οποιασδήποτε διακριτική μεταχείρισης ει βάρο των φίλων. Από τη δική μα την πλευρά είναι σαφέ. Δεν θα κάνουμε ποτέ κανένα βήμα επαναχώρηση στην προάσπιση των δικαιωμάτων και τη ισότητα. Κύριε Πιτέλα, σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Θα τα μεταφέρω ως Προεδρεύων στον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη. Ζήτησε ε, επίσης το λόγο για point of order ο κύριος Κόρβιν Μίκε και έχει το λόγο. You have the floor. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ την ε, αναβολή τη διαδικασία ασυλία τη κυρία Μαρή Λεπέ για του εξή λόγου. Δυστυχώ, αν την ψηφίσουμε τώρα, θα πάρει 100.000 ψήφου παραπάνω. Και έτσι θα κερδίσει και τι προεδρικέ εκλογέ. Θα συμβάλλουμε δηλαδή στη νίκη τη στι γαλλικέ προεδρικέ εκλογέ. Γι' αυτό ζητώ να αναβληθεί η άρση της ασυλίας, γιατί εμείς με τον τρόπο αυτό παρεμβαίνουμε στην εκλογική διαδικασία για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ευχαριστώ. Κύριε Κόρβιν και υπέθετα ότι θα είχατε κάτι να πείτε για όσα ανέφερε ο κύριο Πιτέλα. Πρωτοτυπήσατε. Θε, θέλω να πω ότι με βάση τον κανονισμό σε ό,τι αφορά στο αιτήμα σας, με βάση τον κανονισμό άρθρο 180 παράγραφος 1, οι αιτήσει για την άρση της ασυλίας οποιοδήποτε ευρωβουλευτή γίνονται με ανάταση της χειρός, όχι με ονομαστική ψηφοφορία. Ε, το λόγο έχει ζητήσει επίσης για point of order ο κύριος Γούλφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βάσει το άρθρο 188 και το άρθρο 44 και τη Επιτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων, θέλω να θέσω την κατεπίγουσα υπόθεση του Άλεξ Ανταμέσκου, Γερμανού πολίτη που κατοικεί στο Λονδίνο και ο οποίος έχει υποστεί έχει μάλλον εναντίον του ένταλμα σύλληψη από, τη Ρουμανική, από τις Ρουμανικές Αρχές και τη Ρουμανική Αστυνομία. Ο πατέρας του κ. Ταβέσκου έχει συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες, έχει χάσει τη ζωή του στη φυλακή και η σύζυγός του έγινε απόπειρα να πελαθεί ε, παρανόμω από τον Ηνωμένο Βασίλειο, από γκάγκστερ. Εδώ λοιπόν δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη να χρησιμοποιείται από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτικέ σκοπιμότητε. Σα παρακαλώ να το θίξετε στο ύψιστο δυνατό επίπεδο και να το θέσετε στην προσοχή του Προέδρου ε, τη Αρμόδια Επιτροπή ε, βάσει των σχετικών άρθρων του κανονισμού. Στο, πριν περάσουμε στι ψηφοφορίε, με χαρά απευθύνω χαιρετισμό στον κύριο Χαμπίμπ Αλμάλκη, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βασιλείου του Μαρόκου και στην αντιπροσωπεία του που τον συνοδεύει, οι οποίοι βρίσκονται στο θεωρείο των επισήμων. Ο κύριος Χαμπίμπ Ελμάλκι και η αντιπροσωπεία του πραγματοποιούν χθε και σήμερα επίσκεψη εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας τιμούν με την παρουσία τους στη σημερινή ψηφοφορία. Τους καλωσορίζω θερμά. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Φεράρα σχετικά με την αίτηση ασυλία, έτσι για την άρση της ασυλίας της Μαρίν Λεπέν. Έχει κατατεθεί πρόταση από τον κύριο Κόρβιν, Μίκε για την αναβολή της σχετικής ψηφοφορίας.